για την υβριδοποίηση ε, είναι εντάξει και οπότε δεν μπορούν να ε, έχουν ανετικές συνέπειες στην επικονίαση στη φύση. Για να δούμε τι είναι αυτή η τεχνική πριν ε, μπούμε σε αυτό το χωρό των ανακοινώσεων. Ο κύριος Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κάθε τεχνολογία και κάθε κοινοτομία είναι πρόσδεκτη. Αρκεί όμως να εμπίπτει στο πλαίσιο των κοινών αξιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος Συμβουλίου. Όταν επεξεργαζόμαστε και τροποποιούμε έμβρια, γαμέτες και εν γέννη την ανθρώπινη βλαστική σειρά, τότε πραγματικά οδηγούμαστε σε επιπτώσεις οι οποίες μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνες και για τις επόμενες, τις επερχόμενες γενναίες. Και βέβαια αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και εν γέννη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διεθνής απαγόρευση όσον αφορά την τροποποίηση των γενετικών κυτάρων του ανθρώπου. Τάσομαι υπέρα τον όσων λέγονται στο προφορικό ερώτημα, άκουσα και την κυρία Γιούροβα και θέτω ένα ακόμα ερώτημα. Ποια είναι η αποψή σα σε σχέση με το κινέζικο αυτό πείραμα, ότι όπω ακούσαμε, ενδεχομένω να μην έλαβε χώρα, δεν επαληθεύτηκαν τα πορίσματά του. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και οι Κινέζοι επιστήμονες να ακολουθήσουν τους διεθνείς κανόνες. Κυρία Καπεθόν Ρουίζ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλες επιστημονικές πρόοδοι πάντα ε, γέννησαν πολλές συζητήσεις διοντολογικού χαρακτήρα και ακριβώς αυτή είναι και ε, η κόκκινη γραμμή, η διοντολογία, έτσι ώστε η επιστήμη να είναι ποιοτική. Τώρα θα παραγγέλνουμε έμβρια και θα τα σχεδιάζουμε ε, απαράδεκτο επιστημονικά. Και βεβαίως θα πρέπει να το διαχωρίσουμε από τη γενετική θεραπεία ε, για ορισμένες ε, ασθένειες, ακόμα και τα βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούνται σήμερα στην θεραπεία κάποιων καρκίνων. Δεν θα πρέπει να μπλοκάρουμε τις ευκαιρίες, γιατί αύριο ε, η γενετική θα μας δίνει πολλές νέες ευκαιρίες. Αυτό χρειαζόμαστε συζήτηση για το πλαίσιο, το δεντολογικό, το ρυθμιστικό, το κανονιστικό ε, της νέας αυτής ε, ευκαιρίας του νέου κλάδου που πραγματικά ανοίγει πολλές προοπτικές και ελπιδοφόρες. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Κινέζος αυτός επιστήμονας που ισχυρίστηκε ότι ε, μπορεί να φτιάξει γενετικά τροποποιημένο έμβριο είναι απαράδεκτη. Ε, δεν επιτρέπεται παρέμβαση στην ανθρώπινη βλαστική σειρά. Ε, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, δεοντολογικό και εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να ε, διατρανώσουμε ότι είναι απαράδεκτα. Ε, αυτά τα πράγματα. Η ε, επιστήμη θα πρέπει να μας διευκολύνει να κατανοούμε τον κόσμο που μας περιβάλλει και την ανθρώπινη φύση. Αλλά και οι έρευνες θα πρέπει να σέβονται ε, κάποια πλαίσια. Ναι, να καταπολεμούμε τις ασθένειες, αλλά δεν μπορούμε να δεχόμαστε οτιδήποτε. Ό,τι είναι τεχνολογικά και τεχνικά δυνατό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται κιόλας. Ε, δεν μπορούμε να ε, τροποποιούμε ε, τη βλαστική σειρά και τους γαμέτες, γιατί αυτές οι τροποποιήσεις μεταδίδονται στις επόμενες γενναίες. Δεν μπορούμε να παραγγέλνουμε παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα καταδικάσει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Μοργάνο, για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο συνάδελφο Μιλόζατσικ, καθώ επίση και διάφοροι προλαλήσαντε. Αν τελικά επιβεβαιωθεί το πείρημα αυτό του Κινέζου επιστήμονα, ο οποίο τροποποίησε το ανθρώπινο γονιδίωμα, Σαφώς τότε έχουμε μια παραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται εδώ πέρα σημαντικά ερωτήματα επιστημονικής, κοινωνικής και διοντολογικής φύσης. Η ιατρική και η βιολογική έρευνα σαφώς έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να σημειωθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών και στη μείωση της ανθρώπινης οδύνης. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε την απαραίτητη διάκριση ανάμεσα στην τροποποίηση του γονιδιώματος των σημαντικών κιτάρων και την τροποποίηση της ανθρώπινης βλαστικής σειράς. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το τελευταίο, ακόμα και όταν γίνεται ακούσια, μπορεί να οδηγήσει σε κληρονομήσιμες επικίνδυνες επιπτώσεις, οι οποίες θα περάσουν και στις επόμενες γενές Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σαφώς και στα πλαίσια ακόμα της διεθνούς επιστημονικής έρευνας να τονίσει για μία ακόμη φορά ότι υπάρχουν συγκεκριμένε αρχέ, συγκεκριμένε κόκκινες γραμμές, τις οποίες δεν μπορούμε να υπερβούμε σε καμία περίπτωση. Διακόπτη Πρόεδρος, έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Σα δω συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιποι να πάρουν το λόγο. Η κυρία Γιούροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τις απόψεις σας για αυτό το ιδιαίτερα λεπτό από επιστημονικής και από άποψης θέμα. Όπως είπα και από την αρχή, θα συνεχίσουμε να διαρευνούμε το θέμα, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα επανέλθει στην επικαιρότητα στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστούμε. Τέλος, ο κύριος Τσάμπα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που θίξατε αυτό το ζήτημα. Το Συμβούλιο ε, σημειώνει τα ερωτήματά σας ε, και τις απόψεις σας και σας διαβεβαιώ ότι θα παραμείνει υψηλά ε, στην ατζέντα μας. Σας ευχαριστώ και πάλι την προσοχή σας. Ωραία, συνάδελφοι, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής συζήτησης. Η επόμενη συνεδρίαση είναι, θα αρχίσει στις 9 το πρωί και θα είμαι εδώ και πάλι ω Πρόεδρο. Ελπίζω να είστε και εσεί. Μπορείτε να βρείτε την ημερήσια διάταξη στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Πέρα συνεδρίαση.